Ε, για αυτά τα θέματα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε η πράσινη συμφωνία μας να είναι και γαλάζια. Γιατί όπως ξέρετε το πράσινο δεν υπάρχει χωρίς το γαλάζιο. Χωρίς το γαλάζιο είναι μόνο κίτρινο. Εγώ θα συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο για να υλοποιήσουμε την Πράσινη Συμφωνία, για να διαμορφώσουμε μια φιλόδοξη στρατηγική βιοπικλότητα για το 2030 τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να προετοιμάσουμε μια επιτυχή ε, κοπ στο Κουνμίνγκ τον Οκτώβριο και αναμένω το ψήφισμα που θα υιοθετήσετε αύριο θα μας καθοδηγήσει για να ολοκληρώσουμε και να υιοθετήσουμε τη στρατηγική βιοποικιλότητα τη επόμενη εβδομάδες. Σα ευχαριστώ ξανά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σινκεβίσιο, κύριε Επίτροπε. Ε, Θα έχουμε τώρα ε, την ψηφοφορία αύριο. Πάμε τώρα στην εκθέση του συναδέλφου για αφορά τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δημοσιολαβητή του 2018. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όπως συνηθίστε μπορείτε να δηλώσετε ότι θέλετε να μιλήσετε με το ηλεκτρονικό σύστημα ε, και το ίδιο και για τη γαλαζιά κάρτα. Για να ξεκινήσουμε θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον εισηγητή, τον κύριο Γιάρια, τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη βδομάδα συζητήσαμε εντατικά ότι πρέπει να στραφούν περισσότερο στους πολίτες ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θέλουμε να υπάρχει μια επαφή με τους πολίτες, ώστε αυτοί να μπορούν να συναποφασίζουν πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα προχωρήσει για τον εκδημοκρατισμό, τη διαφάνεια. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά. Αλλά συνάδελφοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή έχουμε έναν θεσμό ο οποίος βρίσκεται κοντά στον πολίτη. Πιο κοντά στον πολίτη. Ε, σχεδόν περισσότερο δεν γίνεται, θα έλεγε κανείς. Με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μπορεί να έρθει ένας πολίτης απευθείας σε επαφή να βοηθήσει να αποφασιστούν πράγματα, να στραφεί σε αυτόν. Ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής είναι εκεί για τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες και όχι για το Συμβούλιο, ούτε την Κομισιόν, ούτε το Κοινοβούλιο. Τι σημαίνει Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής, σημαίνει αυτό ότι μερικές φορές πρέπει να συζητήσει με την Κομισιόν, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, και μερικές φορές ε, πρέπει να συνεργαστεί στενά με αυτούς. Και θέλω να συγχαρώ για την εργασία της στην Εμίλια Ράιλι, τη Δημεσολαβήτρια, για, τις εργασίες, για την εργασία της ε, ε, που καταφέρει να κάνει αυτό το σπαγκάτο, αυτή την επαφή προς όφελος των πολιτών. Σκοπός είναι να παρέχεται ποιοτική υπηρεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιωθεί αυτή η υπηρεσία προς τους πολίτες. Και θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Εμίλια Ωραίλη ε, για θέματα διαφάνειας. Έχει την ε, ε, υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Στο Συμβούλιο δεν ήταν τόσο σύμφωνο με αυτήν, αλλά το έγγραφο του Συμβουλίου είναι ύψη τη σημασίας και θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και από το Συμβούλιο. Αυτό απαιτούμε. Η νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, θα πρέπει να είναι πιο διαφανής, πιο ανοιχτή και πρέπει να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες. Δεν μπορεί ο ένας ε, συνομοθέτης ε, να λειτουργεί ως διπλωματικό φόρουμ. Σύμφωνα με τις συνθήκες θα πρέπει να μπορεί να τηρεί τις ε, μεθόδους εργασίας του στα επίπεδα μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Οπότε ευχαριστώ και τους συνεργάτες για την έκθεση αυτή. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Πιστεύω ότι ετοιμάσαμε μια καλή έκθεση. Μεριμνήσαμε ώστε να αποπολιτικοποιηθεί η συζήτηση, να γίνει πιο ευρεία και στην Επιτροπή Αναφορών ε, έλαβε 28 ε, υπέρ ε, και εγκρίθηκε έτσι στην Επιτροπή Αναφορών και αυτό είναι καλό σημάδι ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ εμάς ε, και της διαμεσολαβήτριας και ελπίζω και να συνεχιστεί το ίδιο και από τη φετινή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γιάρ. Τώρα δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Δημοσιολαβήτρια, την κυρία Ορέλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ κυρία Γιάρ. ευχαριστώ και τους και για τον κόπο σας στην έκθεση αυτή. Πάντοτε είναι ευχαριστησή σα προσφέρουν τη έκθεση, αλλά φέτο έχει ιδιαίτερη σημασία η παρουσίαση, διότι είναι νέο το Κοινοβούλιο, νέα θετή από όλου, καινούριου βουλευτέ και πριν από έναν μήνα ε, δείξατε την ε, εμπιστοσύνη σα, γιατί μου με, με, επιλέξατε και με δεύτερη θητεία. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σα και θα προσπαθήσω να την επιβεβαιώσω. Επίσης, ευχαριστώ τον Επίτροπο Σέχοβιτς που ήρθε διότι είναι αρχή της ε, διαδρομής αυτής της θητείας Επιτροπή. Επιτροπής. Εύχομαι καλή επιτυχία για όλα τα καλά που κάνετε για την Ευρώπη και όχι μόνο. Εγώ είμαι η γέφυρα μεταξύ των πολιτών και τη Δίκη Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποια παράπονα έρχονται αυτά από φυσικά πρόσωπα, από την κοινότητα των πολιτών, από νομικά πρόσωπα, από δημοσιογράφου, αλλά πολλέ φορέ και από ευρωβουλευτές. Και εμεί επικαλούμεθα στην ανάλυση μας όχι μόνο το κοινοτικό δίκαιο, αλλά και τις αρχές της χρηστής διοίκησης και θέλουμε να υπάρχει μια δίκαιη μεταχείριση προς τους πολίτες, γιατί πολλές φορές ε, ε, πνίγονται από την τεχνική φύση, από την γραφειοκρατική φύση της Δίκης Ένωσης. Εμείς δεν είμαστε δικηγόροι. Προσπαθούμε όμως να εξισορροπήσουμε από τη μία μεριά τον πολλέ φορέ ε, αδύναμο καταγγέλλοντα και από την άλλη μέρα τη περιμπανή χειριδίκηση. Το 2018 είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των καταγγελιών και αυτό συνεχίστηκε και το 2019. Αυτό όχι επειδή τα θεσμικά όργανα ε, κατέβασαν τον πύχη, αλλά όλα είναι και περισσότεροι, έμαθαν για τη δική μας υπηρεσία, για το τι έχουμε πετύχει, τι μπορούμε να πετύχουμε και ευχαριστώ τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις υπηρεσίες για τη συνεργασία τους. Σε όλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων που διεκπαιρεώσαμε έγιναν με σημαντική στενή συνεργασία με τη διοίκηση και αυτό θα πρέπει να τον αναγνωρίσω. Ναι, αναδεικνύω τα προβλήματα γιατί αυτό είναι ο ρόλος μου. Επίσης όμως ε, επισημένο την, ε, την ευσυνείδητη δουλειά όλων των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ε, προσπαθούμε όλα αυτά να γίνουν και να τα διαδώσουμε παντού σε όλους τις διοικήσεις. Οπότε είχαμε την λογοτοδοσία, είχαμε διαφάνεια, ε, αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της ύλη που εκπαιδεύσαμε. Το 18 επίσης ε, χρησιμοποίησα κάτι που δεν το τόσο συχνά. Δηλαδή το να υποβάλω μια ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επρόκειτο για την δεύτερη φορά που το έκανα αυτό, από τότε που πρώτο εξελέγην Το 13 απευθύνθηκα σε εσά και είπα ότι αυτή η αρμοδιότητα πρέπει να ασκείται πάρα πολύ σπάνια σε πολύ σοβαρέ περιπτώσει, όταν ένα θεσμικό όργανο δεν ε, πράττει σύμφωνα με τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί. Και έγινε κάποια έρευνα όσον αφορά την λογοδοσία για το Συμβούλιο. Και αυτό έγινε γιατί επισημάθηκε στην νομοθετική διαδικασία έλλειψη διαφάνεια όσον αφορά το νομοπαρασκευαστικό έργο για το κοινοτικό δίκαιο, γιατί ο κόσμο δικαιούται να ξέρει τι κάνουν οι κυβερνήσει όσον αφορά την διαμόρφωση, τη θέσπιση τη νομοθεσία. Πάντω ε, ε, έγινε ε, κάτι το οποίο σήμαινε ότι οι υπουργοί κρύβανε το πώς θεσπίζουν νόμους που επηρεάζουν τους δικούς τους πολίτες. Ε, οπότε τελικά έκανα κάποιες συστάσεις, αντιστάθηκαν κάποια κράτη-μέλη, αλλά όλο ένα περισσότεροι στο Συμβούλιο δημόσια τοποθετήθηκαν υπέρ των μεταβολών που πρότεινα. Τώρα έχουμε 10 κράτη-μέλη. Ελπίζω και αυτή η Προεδρία, αλλά και η επόμενη η Γερμανική, θα πάρει τη σκητάλη για αυτό το θέμα της δημοκρατίας ε, και της ε, νομιμότητας στην κοινοτική νομοθεσία. Εμείς έχουμε 96 γραφεία σε 36 χώρες της Ευρώπης και ε, επίσης συνεργάζεται μαζί μας και η Επιτροπή των Αναφορών. Το 2018 είχαμε μια διάσκεψη τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες. Ο βασικός ομιλητής ο Μισελ Μπαρνιέ και ευχαριστώ πάρα πολύ το Κοινοβούλιο βοήθησε με επαγγελματικό τρόπο και πέτυχε αυτή η εκδήλωση. με κύριοι βουλευτές, στην αρχή της θητείας μου είναι σημαντικό να δούμε τι ρόλο θα διαδραματίσουμε σε σχέση με την αρχιτεκτονική της Ένωσης με ορίζοντα το 2020 και πέρα από αυτό. Η Κομισιόν είναι ένα όργανο γεωπολιτικού χαρακτήρα, μετανάστευση, εξωτερική πολιτική, άμυνα, κλιματική αλλαγή, μαζί με διάφορες υπηρεσίες κοινοτικέ που επίσης θα εποπτεύσουν αυτό το έργο το Κοινοβούλιο. Πρόκειται βέβαια να ασκήσει δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και την υπηρεσία της Διαμεσολαβήτριας. Αυτά τα κάνουμε όσο πιο πρακτικά γίνεται και θέλουμε να δούμε τι γίνεται με το συντονισμό του επαναπατρισμού, έχουμε την, την ΕΑΣΟ για τους ετούντες άσυλο στα ελληνικά νησιά, έχουμε την υπηρεσία άμυνας για να δούμε τι τεχνολογία πρέπει να υπάρχει για τον 21ο αιώνα. Αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θα πρέπει και η δική μας υπηρεσία να προσαρμοστεί για να ε, ευθυγραμμιστούμε αυτούς τους ρυθμούς. Όμως, έχουμε λιγότερες από 70 θέσεις υπαλλήλων και έχουμε όλο ένα και περισσότερες καταγγελίες, ύψη, αριθμή ρεκόρ, όλο ένα και πιο περίπλοκη και το Κοινοβουλίο έχει δει στη διάρκεια του προπολογισμού το πόσο μας λείπουν οι πόροι και συνεχώς έχουμε αναθεώρηση του καταστατικού τη Υπηρεσία μας. Οπότε θα πρέπει σφαιρικά να βλέπετε το πρόβλημα και εσείς και σε συνεργασμό με Κομισιόν και Συμβούλιο και να βρείτε κάποια λύση. Διότι είναι προς το συμφέρον όλων η υπηρεσία μας να είναι πλήρως εξοπλισμένη με ό,τι πώς χρειάζεται για τον επόμενο, μάλλον για τον 21ο αιώνα. Οπότε θα πρέπει να φυγαμιστούμε με τις συνθήκες, με τι προσδοκίε των Ευρωπαίων και σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η γεωπολιτική του κόσμου μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ορέλη. Εκ μέρους της Κομισιόν ακολουθεί ο Επίτροπος κ. Σεφτσοβίτς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Κύριε Διαμεσολαβήτρια, πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα και που έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2019, όπως επίσης και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον κύριο Πίτερ Γιάρε, συντονιστή τον εισηγητή συγγνώμη και τους συντονιστές που εμπλάκηκαν στο έργο αυτό. Η έκθεση αυτή, όπως κάθε χρόνο, προσφέρει ε, σε όλους τους θεσμούς, τις υπηρεσίες, τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα τα οποία θεωρεί ότι είναι σημαντικά. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να έχει καλή διαχείριση στις σχέσεις με τους πολίτες, ε, τις οργανώσεις, ε, τους θεσμούς εθνικούς κλπ. Και δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα της σχέσης αυτής. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσφέρει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες της με λογοδοσία, με επάρκεια και με διαφάνεια και προσπαθεί τα δικαιώματα του πολίτη για την χρηστή δίκηση να τα βάζει στην πρώτη γραμμή. Η συνεργασία λοιπόν με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή είναι στοιχείο κλειδί. Μάλιστα εφόσον τα δύο τρίτα, δηλαδή 285 περιπτώσεις, είχαν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν ξέρουμε ότι εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τον πολίτη. Τα τρία τέταρτα των προτάσεων αφορούσαν τέτοια θέματα. Προτάσεις για λύσεις, για βελτιώσεις ή συστάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συστάσεις, οι προτάσεις για λύσεις από πλευράς του Διαμεσολαβητή οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα ακολουθήσει. Και γι' αυτό τελικά μόνο 6% των ερευνών καταλήγουν να διαπιστώνουν κακή διαχείριση. Δηλαδή, αφού με δέος επιμέλεια ερευνήσει τα θέματα ο θεσμός του διαμεσολαβητή δεν καταλήγει σε συμπεράσματα και κακή διαχείριση από πλευρά της Επιτροπής, είτε γιατί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, είτε γιατί έχουμε καταλήξει σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη συνέχεια. Τα υψηλά πρότυπα πάντως είναι κάτι που τονίζει η διαμεσολαβήτρια όταν να μιλάει για χρηστή δίκηση. Το 2019 αναγνώρισε με πρωτοβουλίες της ότι υπήρξε θετικός αντίκτυπος στις ζωές των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μόνο ε, με μείωση της ρήπανσης από τα πλαστικά, για παράδειγμα, για την ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτό το θέμα. Υπήρξαν ε, διάφορες επιτυχίες σε διάφορες κατηγορίες. Συνεχίζει να δείχνει το δρόμο πάντως ο θεσμός του Ευρωπαίου Λεβητή για να βελτιώνονται οι διοικητικές πρακτικές. Εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίσει την επικοδομητική σχέση που είχε μέχρι τώρα υπέρ του συμφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων. Αξιότιμε Πρόεδρε, προσβλέπω στη συζήτηση με τους ευρωβουλευτές και σας ευχαριστώ και τον προτέρων για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ, κύριε Σεφτσοβιτς. Τώρα δίνουμε το λόγο στον συνάδελφο Τέρες για δύο λεπτά. Αξιότιμε κύριε Πίτροπε, κύριε Ωράιλη, ως σκιώδης συζητητή, μπορώ να σας πω ότι Είναι εύκολο να συντάσει κανεί μια έκθεση δραστηριότητα όταν αυτό που τη συντάσει υπήρξε εξαιρετικά δραστήριο και εξαιρετικά επαγγελματία στη δουλειά του. Ο Σκιώδη για του σοσιαλιστέ όσον αφορά τι δραστηριότητε τη κυρία Σοραϊλή το 2018 εντυπωσιάστηκα από τον επαγγελματισμό, το θάρρο και την αφοσίωση τη κυρία Οραελή καθώς υπεράσπιζε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στη σχέση τους με τα διαφορά θεσμικά όργανα. Το, αυτό δείχνει, αποδεικνύει και η επανεκλογή τη ω διαμεσολαβήτρια. Η διαφάνεια, η λογοδοσία των Ευρωπαίων αξιωματούχων, η πρόσβαση στα έγγραφα και στι πληροφορίε ήταν το μίσο, όπου δραστηριοποιήθηκε έντονα η κυρία Οράιλη και κατάφερε να βρει σωστέ λύσει. Σε αυτά τα θέματα έχουμε προτάσει ε, για υψηλό επίπεδο διαφάνεια σε όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφάνεια είναι βασική συνιστόσα του κράτου δικαίου και θα ήθελα να συστήσω στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προτάσεις της κυρίας Οράιλη στα θέματα αυτά σε όλο. Τη διάρκεια του 2018 απέδειξε θάρρος και αποφασιστικότητα η κυρία Οράιλη κατά του status quo απέδειξε ότι στο υψηλότερο επίπεδο της Επιτροπής Γιουνκέρ υπήρχαν περιπτώσεις ε, σοβαρών παραβιάσεων των κανόνων όπως ε, στην εκλογή του κυρίου Σελμάιερ μετά από τις ε, ρουμανικές εκλογές κάτι τέτοιο θα το αναφέραμε κάτι τέτοιο ως ε, ενεργό διαφθορά και οι υπεύθυνοι θα ε, διώκονταν δικαστικά. Χαίρομαι σήμερα που έχουμε εδώ έναν επίτροπο να είναι παρόν σε αυτή τη συζήτηση, αλλά διάφοροι αξιωματούχοι της ε, Κομισιόν κάνουν κήρυγμα για το κράτος δικαίου και για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε διάφορα κράτη-μέλη, ενώ παραβιάζουν τους κανόνες οι ίδιοι, όπως έκανε η Επιτροπή Γιούνκερ. Θα ήθελα η κυρία Οράλη λοιπόν ε, να την ενθαρρύνουμε να δείξει την ίδια αφοσίωση που έχει δείξει μέχρι σήμερα για την υπεράσπιση των συμφερόντων ε, των πολιτών. Και εμείς ως μέλη της Επιτροπής ε, Αναφορών και του Κοινοβουλίου αυτού υποσχόμαστε ότι θα έχετε την υποστήριξη μας. Καλή δουλειά, καλή τύχη. Ευχαριστούμε κύριε Τερέσα. Τώρα η κυρία Τόμ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μην επαναλάβω ότι προελέχθη θα ήθελα, αλλά δεν έχω το χρόνο, οπότε δεν θα το πράξω. Ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά και συνετήρια την επανεκλογή. πάντω. διαπιστώθηκαν κάποια διαδικαστικά προβλήματα από αυτές τι ε, εκλογέ. Θα πρέπει η Επιτροπή των Αναφορών να μεταβάλει την διαδικασία της εκλογής. Να είναι τα πράγματα όπως αρμόζουν σε διαμεσολαβητή. Διάφανα. Είχαμε κάποια προεκλογική καμπάνια εν μέρη βρώμικη και χρειάζονται και κάποιες προθεσμίες, κάποια χρονικά πλαίσια. Να μην στριμώχνουμε και τα χλωρά και τα ξερά. Συμφωνώ με αυτά που είπατε ε, για το μέλλον, οι συναδελφοί από το ΕΛΚ και από τους σοσιαλδημοκράτες. Πάντως, για την χρηστή διοίκηση θα πρέπει να φροντίσουμε. Και είναι και το θέμα το πώς ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν έχουμε κάποιες καταγγελίες για κάποιες παραβάσεις, για κάποιες παρατυπίες. Όταν απευθύνεται στα κράτη-μέλη, για αν υπάρχει παρέμβαση του κοινωνικού δικαίου, πολλές φορές δίνεται μια απάντηση που ικανοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε και εμάς μας λέει η Κομισιόν ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό του πολίτη που δίνει μια ανήση μάχη με την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Και για το e-pilot θα πρέπει κάτι να δούμε. Οπότε υπάρχουν κάποιε παρατυπίε, δεν υπάρχει διαφάνεια, τα σχετικά έγγραφα, οι φάκελοι πολλέ φορέ. δεν είναι προσβάσιμοι στον κόσμο. Αυτό είναι πρόβλημα. Θέλουμε πιο δυναμική ενεργητική ε, στάση. Φυσικά και θα συνεργαστούμε με τη Δημεσολαβήτρια για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Τόμ. Κύριος Λεμπρετών για δύο λεπτά. Merci, monsieur. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα ηθικής όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί τα θεσμικά τη όργανα ε, παραβιάζουν ακόμα και του πιο στοιχειώδεις κανόνε, όπω για παράδειγμα η Επιτροπή των Βρυξελών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπω αποδεικνύει και η έκθεση του 2018 τη Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η οποία σελίδα 9 καταγγέλει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε τον γενικό της γραμματέα, τον ε, Γερμανό Μαχτελμάγερ, και καταγγέλει συγκεκριμένα τέσσερις περιπτώσεις κακής διοίκησης, μεταξύ άλλων ε, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να προχωρήσει σε αυτόν τον ορισμό, χωρίς να υπάρχει αυτή η έκτακτη ανάγκη. Έτσι λοιπόν αυτά τα πράγματα έπρεπε να προχωρήσουν, Πήγαν στην νομική επιτροπή, αλλά πέρασαν 16 μήνες μέχρι να δοθεί κάποια συνέχεια και να απαλλαγούμε από τον κύριο Σελμάγερ. Ζήτησε επίσης μια συγκεκριμένη διαδικασία για τον ορισμό του Γενικού Γραμματέα. Δυστυχώ όμως στην έκθεσή της λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να δημιουργήσει μια τέτοια διαδικασία. Έλλειψη διαφάνειας, συνεπώς. Η διαμεσολαβήτρια επίσης μιλάει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για τον πρόεδρό της, τον κύριο Ντράγκη, ε, τον οποίο καταγγέλει ότι δημιούργησε την ομάδα των 30, ένα ιδιωτικό σώμα που συμμετέχουν οι επικεφαλείς διάφορων ιδιωτικών τραπεζών. Ο Ντράγκη παραμένει μέλος της ομάδας αυτής και καταλήγει στο συμπέρασμα με ιδιαίτερη ανησυχία ότι αυτό οδηγεί σε αμφιβολίες όσον αφορά την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με τα λόμπι συμφερόντων. Είναι πράγματα που και εγώ καταγγέλω συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρκετή διαφάνεια ούτε ηθική. Ευχαριστούμε κύριε Λεμπρετόν για ένα λεπτό ο συνάδελφος Λοτόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ωραίλη. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τη Δημοσολαβήτρια και για την επανεκλογή της. Αυτή είναι η καλύτερη επιβεβαίωση της ποιότητας της δουλειάς σας μέχρι στιγμής. Η έκθεση για το 2018 επίσης ε, αποτελεί απόδειξη της καλής δουλειάς που κάνετε. Το ECR υποστηρίζει την έκθεση αυτή. Αλλά η αρχή μιας νέας θητείας είναι μια καλή στιγμή για να μιλήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να ρίξετε μια στενότερη μάτια στην έλλειψη σαφήνειας και διαφάνειας στου τριλόγους όπως ονομάζονται γιατί αυτή η διαδικασία έχει αποτελέσει πλέον ανέκδοτο ε, δεν είναι όπω θα έπρεπε το βλέπουμε στο πλαίσιο τη δικής μας δουλειά. Ε, για τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα όπου και εγώ είχα την ευχαριστήση να συμμετέχω υπάρχει έλλειψη διαφάνεια από την αρχή ε, της δημιουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Είμαι πεπισμένος ότι η Δημοσιολαβήτρια θα πρέπει να το κοιτάξει και αυτό με μεγαλύτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Σλοτόφσκι, ακολουθεί για ένα μισή λεπτό ο συνάδελφος Γεωργούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι τελευταίες εκλογές ξαναέδειξαν τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λοιπόν επιτακτικό να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα που μα στέλνουν οι λαοί τη ευρώπη και να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να προσπαθήσουμε περισσότερο να προσπαθήσουμε περισσότερο προ την κατεύθυνση τη απόλυτη λογοδοσία και διαφάνεια των θεσμών ώστε να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε κάθε φαινόμενο κακοδιοίκηση και να εξασφαλίσουμε την τήρηση των αρχών του κράτου δικαίου. μόνον έτσι οι πολίτε θα μπορέσουν να πιστούν και να ταχθούν υπέρ τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν αρκεί λοιπόν να ανοίξουμε την πόρτα για να ακολουθήσουν πολλοί αλλά επιβάλλεται να ρίξουμε και άπλετο φω. εν κατακλείδη οι πολίτε θα πρέπει να γίνουν γνώστε και κοινωνοί τη όλη διαδικασία. διαφάνεια δεν είναι οι πολίτε να μπορούν να πληροφορηθούν πλήρω για ό,τι συμβαίνει αλλά να πληροφορηθούν κατά τρόπο εύληπτο και κατανοητό για να μπορέσουν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο τη νομοθέτηση. στον αγώνα αυτό σύμμαχο έχουμε τη διαμεσολαβήτριά μα Έμιλι o'reilly που για ακόμη μια χρονιά υπηρετεί τη θέση αυτή με απόλυτη προσήλωση. Κυρίες και κύριοι της Κομισιόν και του Συμβουλίου, μην την αγνοήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γεωργούλη. Ακολουθεί για ένα μισή λεπτό ο συνάδελφος κύριος Φούρορε. Grazie Presidente. Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Η χρηστή διοίκηση είναι το έργο σε αυτό περιφρονείται Ευχαριστούμε για την έκθεση τον κύριο Γιάρ. Ε, συνολικά συμφωνούμε, εκτός ε, βέβαια από την παραγωγή για την κεντρική τράπεζα, γιατί εκεί υπάρχει το ζήτημα της δημοσιότητας και της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε διάφορα θετικά σημεία από αποτελεσματική δουλειά. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται για την πρόσβαση όμω στα έγγραφα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αναπαροτρία το δικαίωμα των πολιτών. Και σήμερα έχει θεγεί αυτό το δικαίωμα λόγω του κανονισμού 1049. Είναι θέμα που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και Σύμφωνα 100% ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να τροποποιηθεί αυτός ο κανονισμός. Άρα θα πρέπει να έχουμε πιο αυστηρούς ε, κανόνες και να ανέβει ο... Συνάδελφε κύριε φορόρε, έχετε ακόμα χρόνο ομιλίας. Έχετε ακόμα χρόνο ομιλίας, αλλά θα σας παρακαλούσα να μιλάτε λίγο πιο αργά. Υπάρχει κάποιο όριο ταχύτητα εδώ, γιατί αν οι διερμηνείς ε, δεν μπορούν να σας ακολουθούν, είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι πολίτες να καταλάβουν σε όλες τις γλώσσες ό,τι λέτε. you have to use the button. Και τώρα θα, πρέπει να ξαναπατήσετε το κουμπί του μικροφόνου οπότε και εγώ συμφωνώ, έλεγα με το ότι θα πρέπει να γίνει τροποποίηση αυτού του κανονισμού και υπάρχουν βέβαια και κάποια θετικά σημεία εκεί που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνε και πιο αυστηρή διοντολογία για τι συγκρούσει συμφερόντων. Και έτσι θα πρέπει να παρασχεθούν κάποιε εγγύσει όσον αφορά το καθήκον τη ηθική ακυρότητα. Είναι επομένω δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φοντερ Λάιεν για να δείτε την κακοδιοίκηση, να δείτε τις παραβιάσεις ε, της νομοθεσίας όπως έχει γίνει ε, με Μπαρόσο και Ζελμάκη στο παρελθόν. Να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων και άρα χρειάζεται να αναστραφεί αυτή η τάση για να επιστρέψουμε στην χρηστή, ε, στη χρηστή διοίκηση, την ηθική ακαιρεότητα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε συγκεκριμένο χρόνο αγόρευσης εδώ. Δεν έχει νόημα να προβλέπει κανεί πράγματα και μετά, τα γράφει και μετά να τα λέει με διπλή ταχύτητα. Ε, συναδελφοί, είστε νέος στο κοινοβούλιο. Η συνάδελφος Εύη που είναι δίπλα σα, που καθόταν εκεί παλιότερα, ξέρει ακριβώ ότι υπάρχουν και συνάδελφοι Άλλη, παρακαλώ συμβουλέψτε τον συνάδελφο πώ πρέπει να μιλάει όταν έχει συγκεκριμένο χρόνο ομιλία στο μέλλον. Η κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο Ευρωπαίο Δημοσιολαβητής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη δημοκρατία μα, βελτιώνοντα την δίκηση και διασφαλίζοντα την ηθική των θεσμών μα. Και πολύ χάρηκα που Έμιλι Ορέιλι επανεκλέγει. Η Έμιλι αποτελεί ένα παράδειγμα. Είναι κάποιος ο οποίος υποστηρίζει τη διαφάνεια και τη χρηστή δίκηση. Και μάλιστα ε, τη στιγμή που πολλοί από εμάς, πολλές από τις χώρες μας ε, αμφισβητούν πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δικιά μου η χώρα αποχωρεί και χρειάζεται πολύ περισσότερο να φροντίσουμε για αυτή την χρηστή δίκηση. Είναι τελευταία μου ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπώ την βορειοανατολική Αγγλία, την περιφέρειά μου τόσο πολύ αγαπάω. Ήταν προνόμιο για μένα, ήταν τιμή για μένα και ελπίζω κάποια στιγμή κάποιο άλλο να καθίσει αυτή την έδρα να εκπροσωπεί την περιφέρειά μου. Στο μεταξύ, φεύγουμε. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό, την πόλη, την Κάρλα, τον Μάρτ τον και τον Μάλκομ για την αφοσίωσή τους, για το σκληρό τους έργο σε δύσκολες στιγμές όλο το προσωπικό και την Βρετανική Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Αναφορών. Έχω να πω καλή τύχη και καλό βράδυ σε όλους. Thank Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστούμε κύριε Κέρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστούμε κυρία Κερτάν Ντάρλινγκ. Δεν είναι καθήκον μου, αλλά συγκινηθήκατε. Είπατε για τη βόρειο-ανατολική Αγγλία, όπου εκλεγήκατε. Θα σας παρακαλώ να χαιρετήσετε τους πολίτες εκεί, στην περιοχή σας. Για ένα λεπτό, η συνάλφους κυρία Βέντρεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Κυρία Διαμεσολαβήτρια, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για το έργο του. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από περισσότερη διαφάνεια. Έχει υπάρξει πρόοδος ε, στον εμπορικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να δημοσιεύει τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και τι εντολές να τι δημοσιεύει το Συμβούλιο. Τέτοιε βελτιώσει είναι εφικτέ. το έχουμε όλοι υπογραμμίσει και είναι και αναγκαίε. Το Συμβούλιο πιο συγκεκριμένα πρέπει να διασφαλίσει περισσότερη διαφάνεια στη λειτουργία του. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε να υπάρξει συμφωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα για την εφαρμογή ενός μητρώου διαφάνειας που να είναι υποχρεωτικό και νομικά δεσμευτικό για τα λόμπι πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς οι πολίτες. Έτσι θα καταπολεμήσουμε τον ευρωσκεπτικισμό και έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας και να βελτιώσουμε και να προωθήσουμε τη στρατηγική της διαμεσολαβήτριας. Να ξέρετε ότι εγώ το στηρίζω απόλυτα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βεντρέν για ένα μισή λεπτό η κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την διαμεσολαβήτρια την κυρία Ωραϊλή για την επανεκλογή της τη δουλειά της την εκτίμησε ιδιαίτερα το κοινοβούλιο αυτό εκτιμήσαμε επίσης και το είπατε πολύ σωστά εκτιμήσαμε τη δουλειά της το 2018 στην έκθεση που συζητάμε απόψε μια έκθεση που ξανά ζητά όπως είχαμε κάνει και για την προηγούμενη χρονιά να υπάρχει ένα μητρό διαφάνειας επιτέλους υποχρεωτικό νομικά δεσμευτικό ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τα σημαντικά κενά που υπάρχουν όσον αφορά τις δραστηριότητες των λόμπι. Να υπάρχουν και πιο αυστηροί κανόνες ε, για τα λόμπι, ώστε να αποφεύγονται συγκρουσίες συμφερόντων, αλλά και σημαντικές αλλαγές, ώστε όλες οι διαδικασίες λήψης αποφάσεως να γίνουν πραγματικά διαφανείς ε, και να χαρακτηρίζονται από λογοδοσία. Ή εάν η Επιτροπή Βαντερ θέλει να αλλάξει τα πράγματα όσον αφορά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη επιτροπή θα πρέπει να ε, υλοποιήσει αυτά τα αιτήματα. Εγώ διαφωνώ ωστόσο, και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω αρνητικό για αυτή την έκθεση, στην παράγραφο που αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετα από τα πόσα λέει το κείμενο, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να απαγορευτεί τα μέλη της ε, τράπεζας αυτής να ε, συμμετέχουν σε φόρουμ και κλεισμένων των ε, θηρών όπου συμμετέχουν ε, τράπεζε τι οποίε υποπτεύει η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Εύη, ο κύριο Ατζιού Σαλίμπα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ και εγώ την κυρία Ρέλη που επανεκλέγει. Πρόκειται για μια ψήφο εμπιστοσύνη για το θετικό τη έργο προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των Ευρωπαίων πολιτών στο θεσμό. Πολύ χαίρομαι λοιπόν που στην ετήσια έκθεση αναφέρει η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια πολλά πράγματα για τα θέματα ατόμων με αναπηρίες και πώς θα μεταχειρίζεται αυτά το κοινό καθεστώς υγειονομικής ασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σεβόμενο και τον κανονισμό για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Επίσης, Συμφωνώ με τις συστάσεις που έκανε για καλύτερη προσβεσιμότητα στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Πράγματι, χρειάζεται ένα σύστημα τεχνολογίας που να βοηθάει τα άτομα να συμμετέχουν με συγκεκριμένες δοκιμές που είναι προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες. Τέλος, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ορέλη για το καλό σας έργο και για την αφοσίωσή σας. Θα μας λείψετε. Ευχαριστώ κυρία Ατζιουσαλίμπα. Ακολουθεί για ένα λεπτό ο συνάδελφος κύριος Μπενιφέη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ετήσια έκθεση άλλη μια φορά σας ε, συγχαίρει σας και την υπηρεσία σας για το εξαιρετικό έργο σας. Οι Ευρωπαίοι στο πρόσωπό σα έχουν έναν ε, σύμμαχο. Δίνονται αγώνε ούτω ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυνη λειτουργία της διοίκηση, διαφάνειας, αποφάσεις, ε, η ποιότητα της ε, διοίκηση προ τον κόσμο. Οπότε, Έμιλιο Ράλια, σας ευχόμαστε καλό κουράγιο για την καινούργια σας θητεία και θα πρέπει με αποφασιστικότητα να δείτε τα εξής, έχουμε βελτίωση στη λήψη φάσεων στο Συμβουλίο και πάντοτε αποφασιστικά να είσαστε κόντρα στην κακοδίκηση όπως είχε γίνει τότε με τον ορισμό του Σελμάιερ ως Γενικού Γραμματέα στην Κομισιόν. Είχαμε τότε την συνεργασία με τον διαμεσολαβητή για να σταματήσουν να υπάρχουν ε, τέτοιου είδους ε, ε, δωροληψίες και δωροδοκίες και επίση, όσον αφορά και τα στάζ, τα μη ε, ε, αμοιβόμενα στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε κύριε Μπενιφέη. Πάμε στο Κατσδιάι. Συνάδελφε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώ να σας πω ότι συμφωνώ με την έκθεση. Και Υπάρχει και ένα άρθρο το οποίο μπορεί να μην σας φαίνεται τόσο σημαντικό, όμως είναι πολύ σημαντικό. Είναι το άρθρο 47. Εκεί αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ηθική ακεραιότητα, θα πρέπει να υπάρχει αμεροληψία. Ε, μπορεί πολλοί από σας να θεωρείτε ότι αυτό είναι τυπικό Αλλά ξέρετε τώρα στην ε, Τσεχία είναι πολύ επικαιρό το θέμα. Είχε κατηγορηθεί ο δημοσιολαβητής ότι είχε έρθει σε συμπερινία με εισαγγελική αρχή για να καταδικαστεί κάποια συμπολίτες άμεσα σε θάνατο. Αυτά επομένω δεν είναι αντιεπαγγελματικά Γίνεται είναι και θέμα ε, προσωπική ηθική ακυρότητα. Ευχαριστούμε κύριε Ποσπισίλ. Ο κύριος Λόπες Αγγελάρ. Uh, ευχαριστώ. Πρόεδρε Βίλαντ, ευχαριστώ Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς, ευχαριστώ κύριε Ρέλη. Θέλω και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου στις ε, εκτιμήσεις, στις ευχαριστίες στον θεσμό του διαμεσολαβητή και στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και κυρίως να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε άλλα πέντε χρόνια. Δείχνει την εκτίμησή μας στο έργο σας υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας, πρόσβαση στα έγγραφα, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν παρόλο που τα εμποδίζει το Συμβούλιο παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η Επιτροπή Λίμπε, της οποίας είμαι εγώ πρόεδρος. Μένει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει για να διασφαλίσουμε ότι η σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει πια, ότι οι περιστρεφόμενες πόρτες δεν υπάρχουν πια, ότι οι έρευνές σας για διάφορες πρακτικές ορισμένων κλάδων όπως του φαρμακευτικού συνάδουν με την ε, Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα άτομα με αναπηρίες κλπ. κλπ. Όλα αυτά πρέπει να περάσουν και να γίνουν πραγματικά ευρωπαϊκός κανονισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λόπης Αγγελάρ. Κλείνει η διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και τώρα δίνουμε το λόγο στους αρχικούς ομιλητές ε, με την αντίστροφη σειρά. Ξεκινάει ο κύριος Σεφτσοβίτς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κύριε Ρέιλι, Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα όσα είπατε και για τα σχόλιά σας. Ξεκίνησε ο κύριος Γιάρ και όλοι συμφωνήσατε για το εξαιρετικό έργο της κυρίας Ορέιλι. Ε, σχόλια με τα οποία συμφωνεί απόλυτα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω όμως να πω στην κυρία Τόμο ότι αν πρόκειται για παραβιάσεις και τέτοιες διακασίες, ευχαρίστως να συζητήσουμε Έχω πρόσκληση για την Επιτροπή Αναφορών και θα πάω και θα συζητήσουμε μαζί πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Επίσης θέλω να ενημερώσω τους αξιότιμους ευρωβουλευτές ότι ακολουθήσαμε σωστές διαδικασίες και καταλήξαμε να εκλέξουμε ως Γενικό Γραμματέα έναν πάρα πολύ ικανό ε, πρόσωπο που θα είναι σίγουρα εξαιρετικός Γενικός Γραμματέας, τον κύριο Γιώχανσον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί πάντα να πετύχει το καλύτερο δυνατόν επίπεδο χρηστής δίκησης και θα φροντίσουμε όπως λέει και η συνθήκη και η συνθήκη για τα θεμελιώδη δικαιώματα θα φροντίσουμε και εμείς να τα σεβόμαστε πλήρως. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι οργανώσεις με τις οποίες έχουμε σχέσεις Σίγουρα αναμένουν να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται από τη δικιά μας ε, την πλευρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τονίζω επίσης το γεγονός ότι οι καθημερινές μας ανταλλαγές με τη διαμεσολαβήτρια μας βοηθούν να κάνουμε τη δουλειά μας ε, ακόμα καλύτερα καθημερινά και να ακολουθήσουμε ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα. Να μην υπάρχουν ε, διακρίσεις, να είμαστε αμερόληπτοι και να συμμορφωνόμαστε με τόσα και εσείς αναφέρατε στις παρεμβάσεις σας. Το η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για το έργο της Διαμεσολαβήτριας αναφέρει διάφορους τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Πράγματι, τις επόμενες εβδομάδες θα εξετάσουμε το ψήφισμά σας και θα απαντήσουμε σε όλα τα θέματα τα οποία θίγεται εκεί. Θέλω επίσης να αποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ και τον κύριο Κόρμπετ και όλους τους άλλους συναδέρφους από το Ηνωμένο Βασίλειο για την αφοσίωσή τους, για το σκληρό τους έργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και να ξέρετε ότι θα μας λείψετε πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε πίτροπε, κύριε Σεφτσοβιτς. Διαδικαστικό. Uh, Μάρος, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει όσον αφορά τη νέα πράσινη συμφωνία. Για την φτώχεια επίσης. Ήθελα να πω ότι χρειάζεται για την ενεργειακή φτώχεια να διαμορφωθεί, να θεσπιστεί ένα ορισμό σε αυτή τη θητεία. Και πάλι σε ευχαριστώ για τόσα έκανες για τους μη προνομιούχους Ευρωπαίους. Ήταν διαδικαστικό. Δεν ήθελα να διακόψω. Κυρία Ορέλε. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλους σας ευχαριστώ. Είναι πηγή έμπνευσης όλα όσα είπατε, η υποστήριξή σας, οι προτάσεις σας και περιμένω να τα συζητήσουμε περαιτέρω στο μέλλον. Να, πρώτα απ' όλα την κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ. Ε, δεν είναι και πάρα πολύ συχνό ένα Ιρλανδό να στεναχωριέται που φεύγει κάποιο ε, Βρετανό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ναι, αυτό αισθάνομαι. Και σε ευχαριστώ για την συνεργασία, για την υποστήριξη με την υπηρεσία μας γενικότερα τα τελευταία χρόνια του τελευταίους μήνες επίσης εντυπωσιάστηκα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για όλους σας αλλά εσείς συνεχίσατε ε, με επιμέλεια, με ε, πάντου σε όλους τους χώρους ενώ υπήρχαν τόσα άλλα πράγματα που σας αποσπούσαν την προσοχή εύχομαι καλό κουράγιο και θα μας λείψετε. Τώρα, για να δούμε αυτά τα οποία αναφέρατε. Ε, ευχαριστώ για τα όσα κάνατε για να βοηθήσετε το έργο μας γιατί λάβατε υπόψη τα σχετικά με την διαδικασία και τις διατάξεις που διέπουν την εκλογή του Διαμεσολαβητή δεν θα με απασχολήσουν σε πέντε χρόνια αλλά είναι σημαντικό αυτό όσον αφορά τη διαδικασία αυτήν τώρα όσον αφορά την υπόθεση για τον διορισμό του προηγουμένου Γενικού Γραμματέα στην Κομισιόν ε, όντως ε, ε, δεν απεδέχτησαν τις συστάσεις μας αλλά ο αντιπρόεδρο Σεύκοβιτ σας είπε ότι τώρα τα πράγματα γίνανε αλλιώς και ο νέος γενικό γραμματέας διορίστηκε σύμφωνα με όλες μας τις συμβουλές και προτάσεις κατόπιν εκείνης της έρευνας. Κύριε Σλοτόφσκι, είχαμε τους τριμερείς διαλόγους, εκκρεμεί ακόμη το θέμα και θα το ξαναεξετήσουμε. Κύριε Γεωργούλη, όντως η συμμετοχή των πολιτών είναι πολύ σημαντική, για την ε, νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το θέμα της δουλειά μας. Όντως το 1049 είναι ο κανονισμός που πρέπει να τροποποιηθεί και ολοένα και περισσότερα έγγραφα να είναι προσβάσιμα στον κόσμο που υπηρετούμε. Διαφάνεια στο Συμβούλιο βεβαίω έχει γίνει πρόοδος και υπήρχε ένα θέμα που παλιά αυτό ήταν ε, κάτι που συζητούσαν μόνο σε Βρυξέλλες και στα Σβούργα, τώρα το συζητούν όλοι παντού. Και για την Κεντρική Τράπεζα, για όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες στον κόσμο, ώστε να υπάρχει έλεγχος και υποχρέωση λογοδοσίας. Ε, βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα θέματα της τεχνολογίας και στα σοβαρά μάλιστα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα η WAS είπε ότι, θα, ότι έχει κάποιες θέσεις για ε, μαθητεία κάποιων επαμοιβή. Το το είπε ο κύριος Μπενιφέ. Θα πρέπει αυτό να το διερευνήσουμε περισσότερο. Και πάλι ευχαριστώ για τη βοήθειά σας και για την επανεκλογή μου και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε για αυτό το σημαντικό καθήκον. Ευχαριστούμε κύριε Ωρέλη. Το τελευταίο λόγο έχει ο εισηγητής για δύο λεπτά, ο συνάδελφος Γιάρ. Ευχαριστώ. Ε, ήταν εξαιρετική συνεργασία το τελευταίο χρόνο μεταξύ μα με την Επιτροπή Αναφορών και την κυρία Ωραίλη. Πρέπει να πω ο, ότι βέβαια με αυτό δεν είναι όλα εντάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταφέραμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα μαζί. Αυτό είναι βέβαιο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε δεν πρέπει να σταματήσουμε, απομένουν πολλά να γίνουν. Οπότε α ανασκουμποθούμε και στην Επιτροπή Αναφόρων θα σας υποστηρίξουμε για τα πράγματα που έχουμε μπροστά μας όσον αφορά τη διαφάνεια και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Μαζί θα πρέπει να τα οργανώσουμε τα πράγματα. Λυπάμαι ε, που, φεύγουν, ε, που φεύγει και η κυρία Κέρτον Τάρλινγκ από την Επιτροπή μας. Εγώ συντονιστής του ΕΛΚ ε, συνεργάστηκα με κάποιους ε, ε, συντονιστές των σοσιαλιστών. Είναι λάθος η απόφαση, πιστεύω, να φύγει η χώρα σας και λυπάμαι που θα φύγετε κι εσείς, αλλά θα μείνετε μαζί μας και να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας. Αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία, πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Και αυτό θα μας ε, βοηθήσει να έχετε και την πολιτική μας υποστήριξη, κύριε Ράιλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η ψηφοφορία θα γίνει όπως υπόθηκε αύριο. Και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Η μεταρρυθμίση των Γενικών Αρχών Επιτροπολογίας. Δήλωση της Επιτροπής. Και εδώ και ξανά να σας υπενθυμίσω ότι όπως συνηθίζετε με το ηλεκτρονικό σύστημα μπορείτε να εγγραφείτε για να λάβετε το λόγο ή για να χρησιμοποιήσετε την μπλε κάρτα. Οι οδηγίες υπάρχουν στην είσοδο της αίθουσας Ολομέλειας. Ξεκινάμε εξ ονόματος της Επιτροπής, ο Επίτροπος κ. Σεύτσοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα επιφυλάσσομαι από την ευκαιρία αυτή για να συζητήσω μαζί σα στο πλαίσιο τη επιτροπολογία. Η συνθήκη τη Λισαβόνα εισήγαγε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις κατεξουσιοδότηση και τι εκτελεστικέ πράξει. Και έτσι καταλήξαμε και στον κανονισμό για την επιτροπολογία που θέτει του κανόνε για τον έλεγχο των χωρών μελών επί τη άσκηση των ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις εκτελεστικές πράξεις που στέλνει η Κομισιόν στις χώρες μέλη. Επίση, υπάρχει και δικαίωμα ελέγχου κάθε φορά που φαίνεται να υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Επιτροπή. Ο κανονισμός τηρεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι λοιπόν 1.633 εκτελεστικές πράξεις είχαμε και δεν υπήρξε αρνητική άποψη και υπήρξαν 32 περιπτώσεις μη γνωμοδότησης το 2018. Αυτές οι τελευταίες σημαίνει ότι δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά μια εκτελεστική πράξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είτε επειδή είναι αντιφατικέ οι απόψει των χωρών μελών, είτε επειδή καταλήγουν σε αποχή. Σε ειδικέ περιπτώσει, πάντω, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη δική επιτροπή πρεπει να ζητηθει γνωμη δικη επιτροπη οταν δεν έχουμε γνωμοδότηση. Είχαμε θέματα υγείας και ε, πολιτικής επιτοκαταναλωτών. Σε 12 περιπτώσεις όμως η Επιτροπή κατέληξε σε αρνητική γνωμοδότηση ή όχι σε γνωμοδότηση. Είναι πολύ περιορισμένες οι περιπτώσεις που κατέληξαν σε συζητήσεις γιατί ε, πρόκειτο για πολύ ευαίσθητα θέματα για τα γενετικά τροποποιημένα, ε, τρόφιμα και ζωοτροφές ή για θέματα φυτοφαρμάκων. Όταν επίσης η Επιτροπή αυτή καταλήγει ε, σε μη γνωμοδότηση, μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κανονισμός της κομιτολογίας έχει την ε, λογική που λέει ότι εάν υπάρχει άποψη κατά από την Ειδική Επιτροπή δεν προχωράει. Αυτή ήταν μια αρχή της Επιτροπολογίας από την αρχή για να υπάρχει καλή εφαρμογή των κανόνων. Είχαμε 12 λοιπόν εκτελεστικές πράξεις στα θέματα της υγείας και ε, της προστασίας των καταναλωτών και υποχρεώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει στην απόφασή της βάσει ε, συγκεκριμένων στοιχείων. Αυτές οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία στην αρμόδια Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάζεται μερικέ φορέ να πάρει μη δημοφιλεί αποφάσει. Αποφάσισε λοιπόν να προτείνει ω προτεραιότητα η Κομισιόν να αλλάξουν αυτοί οι κανόνε και να υποβληθούν τροπολογίες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δική αυτή επιτροπή, ώστε να υπάρχει λογοδοσία από τι χώρε μέλη κατά τη διάρκεια τη διαδικασία. Πρόκειται για τι εξή τροπολογίε. Πρώτον, υπολογίζεται η ειδική πλειοψηφία που, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ε, τι χώρε που να μην λαμβάνονται υπόψη χώρε που δεν είναι εκεί που κρατάνε αποχή. Δεύτερον, να υπάρξει και δεύτερη παρουσία του θέματος, υποβολή του θέματος όταν είναι προβληματικά τα ζητήματα. Έπειτα, οι εκπρόσωποι των χωρών μελών να ψηφίζουν ανοιχτά, δημόσια, κάτι το οποίο συζητήσαμε και πριν από λίγο, το διαφάνεια. Έπειτα να υπάρχει και δυνατότητα το θέμα να πάει και στο Συμβούλιο για μην δεσμευτική γνωμοδότηση και πολιτική καθοδήγηση. Πού βρισκόμαστε σήμερα? προτείνεται προτείνονται αυτά τα θέματα επειδή δεν υπήρξε πρόοδο τα τελευταία τρία χρόνια. Από το Συμβούλιο δεν υπήρξε στήριξη στην πρόταση αυτή. Από πλευρά του Κοινοβουλίου η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων απλώς γνωμοδότηση παρουσίασε στηρίζοντας την πρότασή μας και όχι έκθεση. Οπότε, Πρόεδρε, χαιρόμαστε για τη σημερινή συζήτηση γιατί μας δίνει την ευκαιρία να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και ρεαλιστικοί αν δεν υπάρξει κάποια κίνηση ώστε να ξεμπλοκάρει ο φάκελος αυτός, δεν πρόκειται να καταφέρουμε πρόοδο σύντομα. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις δικές σας απόψεις για να αποφασίσει πώς να προχωρήσει στα πλαίσια της αξιολόγηση όλων των εκκρεμούντων υποθέσεων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασία τη Επιτροπή για το 2020. Πάντω, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα για να ζητούμε από τι χώρε μέλη να λαμβάνουν τι ευθύνε του στα θέματα τη επιτροπολογία και για να καταλήγουμε σε αποφάσει με τι χώρε μέλη. Αλλά κάποια συγκεκριμένα βήματα για να βελτιωθεί η διαφάνεια τη επιτροπολογία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σώμα, ξέρω. Σύντομα θα ξεκινήσουμε με ένα νέο μητρό <clears throat> σύγχρονο επιτροπολογίας, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων, αλλά να υπάρχει και πιο εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες. Επίσης, θα συνεργαστούμε μαζί σας και με το Συμβούλιο, ώστε τα μη δεσμευτικά κριτήρια τόσο στις κατεξοδότης όσο και στις εκτελεστικές πράξεις που συμφωνήσαμε πέρυσι θα διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί τα κριτήρια για την προετοιμασία νομοθετικών προτάσεων. Εκ παραλίλου, αξιότιμοι προβουλευτέ, πρέπει από κοινού να έχουμε διαπραγματεύσεις για πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον έλεγχο. Έχουμε πετύχει πέρυσι με το πρώτο πακέτο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα κομμάτια του πακέτου. Προσβλέπω λοιπόν στις δικές σας απόψε εδώ, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε ε, στο έργο μας σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας μας για φέτος. Ευχαριστούμε κύριε Πίτρο Σεύτσοβιτς για ένα μισή λεπτό ο συναδελφός Σάιερ. Ε, Νομίζω ότι δεν έχετε ανάψει το μικρόφωνο, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντιπρόεδρο που εκπροσωπεί την Κομισιόν για τα λόγια του. Ήθελα να πω ότι στο τέλος της προηγούμενης θητείας μας έκανε έκπληξη το ότι σημειώθηκε και κάποια πρόοδος όσον αφορά την ε, επανευθυγράμμιση στο τομέα της ετροπολογίας, αλλά σε αυτό το φάκελο δεν έχουμε προχωρήσει. Η Επιτροπή Γιούρη μόλις πρόσθεσε τη διαδικασία να ξεκινήσει να το εξετάζει οι άλλε, η ΑΦΚΟ, η ΕΚΟΝ και άλλε παρέχαν γνωμοδοτήσει για τον προτινόμενο κανονισμό. Αυτέ οι γνωμοδοτήσει υπογραμμίζουν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί το πλαίσιο επιτροπολογία, όπω έχει, επειδή λειτουργεί εντάξει, αλλά συμφωνούν επίση ότι η διαφάνεια πρέπει να βελτιωθεί περισσότερο. Στη Ιουρή επίση εστιαζόμαστε στο ζήτημα αυτό που απαιτούν οι άλλε επιτροπέ, ειδικότερα στην πολιτική διαφάνεια και τη λογοδοσία σε πολλές ε, υποθέσεις σημαντικές σύμφωνα με την σημερινή διαδικασία η απουσία σαφούς θέσης των κρατών μελών η πολιτική ευθύνη για την τελική απόφαση τελικά έχει η Κομισιόν η οποία χωρίς σαφή πολιτική υποστήριξη από τα κράτη-μέλη βρίσκεται σε ανεπιθύμητη θέση. Η μεταρρυθμίση του 2017, όπως παρουσιάστηκε, ήθελε να διορθώσει αυτή την κατάσταση πρέπει να τονίσουμε ότι αντιλαμβανόμενοι το πόση αντίσταση έχουν φέρει τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, το μέλλον αυτής της μεταρρύθμισης είναι εντελώ απρόβλεπτο και μάλλον όχι ιδιαίτερα θετικό. Λυπάμαι που το κομμάτι της πρότασης που προκαλεί αυτή το διαφωνία μεταξύ κρατών μελών επηρεάζει και τις άλλες συστάσεις που κατά τα άλλα είναι πολύτιμες και ε, που θα εξυπηρετούσαν για καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σάιερ. Για δύο λεπτά η κυρία ο κύριος Κόρμπετς ζητά κύριε Σάιερ. Κύριε Σάιερ. Κύριε Σάιερ. Θέλετε μια ερώτηση από τον συνάδελφο Κόρμπετ. Δεν συμφωνείτε ότι έχει ανατεθεί στην Επιτροπή να αποφασίζει όταν δεν μπορεί να συμφωνήσουν τα κρατημέλια. Μιλούμε για εφαρμογή νομοθεσία που έχουμε ψηφίσει, αλλά το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον ΑΒ τρόπο. Δεν είναι παράλογο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τι ευθύνε τη και εκείνη να αποφασίσει. Και τελικά πρόκειται για εκτελεστικό όργανο που λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο. Επομένω η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει και να μην απεκδίεται αυτές τις, τις ευθύνες με αυτή την πρόταση. Σάιερ. Μάλιστα. Όχι, όχι. Δεν είμαι κατά αυτής της λύσης. Πάντως από ό,τι ξέρουμε επί χρόνια έχει κολλήσει το θέμα στο Συμβούλιο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να πιέσουμε, να, να, να προωθήσουμε με ενθουσιασμό αυτό το οποίο είπατε, αλλά πρότεινε ο Επίτροπος να επιδείξουμε φαντασία, ιδίω εκεί που μπορούμε να έχουμε περισσότερε υποχρεώσει λογοδοσία και διαφάνεια. Ιδίω εκεί που μπορεί να υπάρχει συμφωνία. Ευχαριστούμε κύριε Σάγερ. Η κυρία Φόλατ για δύο λεπτά. Αξιότιμη κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, με αυτή τη συζήτηση πρέπει να δούμε δύο βασικές έννοιες, την λογοδοσία των κρατών μελών και τη διαφάνεια για τους λαούς μας. Όπως είπε ήδη ο Επίτροπος, πολιτικά είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Οι άμεσες επιπτώσεις για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών ε, όπως